για την προκειμένη περίπτωση επειδή εγκατέλειψαν ε, το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Επίτροπο. Ολοκληρώνεται τη συζήτηση και προχωρούμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης έκθεση Τσίστερ για την Ευρωπαϊκή τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών, την ΕΝΙΖΑ. Ο εισηγητής έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Κύριε Τσίστερ. Πρόεδρε, επίτροπε, συνάδελφοι. Πρόκειται, μιλάμε για έναν οργανισμό που ασχολείται με την ασφάλεια δικτύων και πληροφοριών. Είναι η τρίτη ή τέταρτη προσπάθεια που κάνουμε για να ορίσουμε το ρόλο, τα καθήκοντα και τους στόχους του οργανισμού αυτού. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την ομάδα σκιωδών εισηγητών, τον κύριο Έλερ ιδίω, για την επικοδομητική βοήθεια στην διαμόρφωση της έκθεσης. Ευχαριστώ επίσης την Επιτροπή για την υποστήριξη και την επικοδομητική προσέγγιση στο την προσπάθειά μας να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα και αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας ε, του οργανισμού αυτού. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης την Ιρλανδική, την Κυπριακή, την Δανική, την Πολωνική και την Ουγγρική Προεδρίες που όλες διαπραγματεύθηκαν το περιεχόμενο του κανονισμού. Και να πω στους συναδέλφους στο Κοινοβούλιο ότι αν δουν το κείμενο του κανονισμού όσο έχει τώρα, θα δουν τη δουλειά μας. Πόσο άλλαξε τον κανονισμό. Ουσιαστικά και σημαντικά τροποποιήσαμε και βελτιώσαμε ελπίζω το κείμενο. Ο οργανισμός τώρα είναι σε καλύτερη θέση για να αντιμετωπίσει το μέλλον του. Το θέμα της ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών είναι πολύ σημαντικό και είναι ζωτικό να έχουμε έναν ευρωπαϊκό οργανισμό σχετικά επανακαθορίσαμε τις αρμοδιότητες, τους στόχους και τα καθήκοντα, όπως σας είπα, του οργανισμού. Εισαγάγαμε ένα βαθμό διαχείρισης μέσω ενό εκτελεστικού γραφείου που πιστεύουμε ότι θα βελτιώσει τη διαχείριση του οργανισμού. Αναθεωρήσαμε τις ε, ευθύνες του Διοικητικού Συμβουλίου και αυξήσαμε την λειτουργικότητα του οργανισμού ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Εκτελεστικό Διευθυντή να υποχρεούνται να έρχονται στο Κοινοβούλιο και να λογοδοτούν ή τέλο πάντων να παρουσιάζουν τι κάνουν. Εισαγάγαμε ρυθμίσει που επιτρέπουν στο Ελεγκτικό Συνέδριο και την Όλαφ να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες για τις δραστηριότητε του οργανισμού, κάτι δε πολύ σημαντικό, δώσαμε, προβλέψαμε να υπάρξει ένα γραφείο του οργανισμού στην υπηρετική Ελλάδα. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, η υπηρεσία του οργανισμού αυτού είναι στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Πανέμορφο μέρος μεν, αλλά λίγο άβολο ως προς τις ε, μεταφορές και τις επικοινωνίες με την υπόλοιπη Ευρώπη. Δώσαμε προθεσμία, θέσαμε προθεσμία 7 ετών, ε, θητεία 7 ετών στον οργανισμό και προβλέψαμε ότι θα γίνει αναθεώρηση της λειτουργίας το 5ο έτος. Πιστεύω ότι με όλα αυτά τα μέτρα θα βελτιώσουμε την προετοιμασία του οργανισμού για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τα θέματα που προκύπτουν από την κυβερνοασφάλεια τα επόμενα έτη. Πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει την Ένωση, θα ενισχύσει την ικανότητα της Ένωσης, ενώ τονίζουμε την ανάγκη μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου φορέα, ενώ δίνουμε ευελιξία στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, κάποια από τα οποία δεν ξέρουμε καν ποια θα είναι. Σας προτείνω λοιπόν να εγκρίνετε την έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Κρούς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αυτός ο κανονισμός αποδεικνύει ότι καλό είναι να μην τα παρατάει κανείς αν θεωρεί ότι αυτό που κάνει είναι εύλογο. Οπότε θεωρώ ότι έχει γίνει πολύ καλή δουλειά χάρη και στην στάση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για να υπάρξει ένας νέος κανονισμός για τον ΕΝΙΣΑ γιατί έτσι θα υπάρχει νέα, αλλαγή, νέα εντολή, συγγνώμη, σαφής για τον οργανισμό αυτό και θέλω να ευχαριστήσω από την καρδιά μου τον κύριο Τσίτσεστερ και τους σκιώδεις του για το φάκελο αυτό. Έχει γίνει πολλή δουλειά και γνωρίζω ότι ο κατάλογος των προεδριών στις οποίες πρέπει να είναι κανείς ευγνώμων είναι αρκετά μακρύς τον ανέφερε ο εισηγητής και αυτό είναι ένα σημάδι που δείχνει ότι αυτό το θέμα έχει απασχολήσει πολλούς και έχει συζητηθεί εις βάθος. Η Κομισιόν θεωρεί ότι είναι ζωτική σημασία να συνεχίσει τη λειτουργία του ΟΕΝΗΣΑ με αποτελεσματικό και λειτουργικό τρόπο. Αυτή ήταν η αρχή και της συζήτηση. Μιλούμε και για την στρατηγική για την κυβερνοασφάλεια που πρόσφατα ξεκίνησε για την Ευρώπη και γι' αυτό χρειαζόμαστε τον ΕΝΙΣΑ. Ο ΕΝΙΣΑ πρέπει να παίξει ε, ρόλο κλειδί έτσι ώστε η Ευρώπη να βελτιώσει την αντίσταση και την ασφάλεια των δικτύων της και των συστημάτων πληροφοριών. Στην αρχή όταν πρωτοειδρύθηκε ο ΕΝΙΣΑ δεν ήταν σαφή τα πράγματα, τώρα όμως είναι απολύτως σαφή. Τον χρειαζόμαστε, τον οργανισμό αυτό και χαίρομαι που μετά από μακροσκελείς συζητήσει. εγώ δεν πιστεύω στην αιώνια ζωή, αλλά καμιά φορά είχα την εντύπωση ότι έπρεπε να έχουμε αιώνια ζωή για να καταλήξουμε στο τέλος αυτής της διαδικασίας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ήταν δύσκολε μερικέ φορέ συζητήσει, αλλά τώρα έχουμε καταλήξει σε μια νέα εντολή. Οπότε τώρα μπορούμε πια να βασιστούμε σε αυτή την επιτυχία που έχουμε με τούτο τον οργανισμό και αυτό συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων και ε, τομείς όπως ε, το, το πανευρωπαϊκό εγχείρημα για την ε, ε, κυβερνοασφάλεια, σχέσεις με τρίτες χώρες, ανάλυση παγκοσμίων απειλών, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε τομείς κλειδιά και βεβαίως η νέα αυτή εντολή θα επιτρέψει στον ΕΝΗΣΑ να παίξει το ρόλο που πρέπει σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των δικτύων και πληροφοριών. Ο ΕΝΗΣΑ λοιπόν θα είναι πιο αποτελεσματικός, θα είναι πιο κοντά σε αυτούς που τον χρησιμοποιούν, είτε είναι τα ευρωπαϊκά όργανα, γιατί εδώ μπορείτε να βασιστείτε στο ότι θα είναι αποτελεσματικός για εσάς, αλλά είτε είναι τα κράτη-μέλη ή οι ιδιωτικές εταιρείες αυτοί που χρησιμοποιούν τον ΕΝΙΣΑ και μπορούν να ωφεληθούν από αυτόν. Τέλος, η Προεδρία έχει επιβεβαιώσει ότι το Συμβούλιο θα υιοθετήσει τον συμφωνημένο ε, ε, συμβιβασμό, οπότε περιμένουμε και εμείς την τελική σας ψηφοφορία αύριο. Κλείνοντας, να πω ότι είμαστε ευγνώμονες. Υπάρχει μέλλον για τον ΕΝΙΣΑ, χρειαζόμαστε τον οργανισμό αυτό Τώρα υπάρχει σαφήνεια και για όσους εργάζονται στον οργανισμό αυτό. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ, Επίτροπε. Δεν βλέπω εδώ την κυρία Χάουγκ. Συνεχίζουμε με τους αγωγητές των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος Έλερ για δύο λεπτά. Για το ΕΛΚ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Αντιπρόεδρε Κρούς, κύριε Τσίτσιστερ, αγαπητοί συνάδελφοι και συνεισηγητές. Ο ΕΝΙΣΑ δεν είναι αυτός ο σκοπός. Ο ΕΝΙΣΑ δεν ε, είναι μια υπηρεσία. Ε, η συζήτηση για τον ΕΝΙΣΑ είχε να κάνει με τις ε, τεράστιες προκλήσεις που έχουμε για την εσωτερική αγορά, για την ελευθερία των πολιτών, για την ελευθερία και την ασφάλεια, της νέας ψηφιακής γενιάς. Αυτό που μπορεί να κάνει και που πρέπει να κάνει ο ΕΝΙΣΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι να έχει την εμπειρογνωμοσύνη, τον συντονισμό, τη συνεργασία, τη συνεργασία και με τα κράτη-μέλη που δεν έχουν φτάσει ακόμα πολύ μακριά σε αυτό το τομέα για να αντιμετωπίσουν τέτοια προβλήματα. Ο ΕΝΙΣΑ είναι ένας λίθος ε, πάνω στον οποίο θα βασιστεί η στρατηγική μας για να προχωρήσει ας πούμε το κέντρο για τη, της Europol για την ασφάλεια ή ένας λίθος πάνω στον οποίο θα βασιστούν οι διάφορες ε, οδηγίες που έχει ήδη υποβάλει η Επίτροπος Κρούς για την κυβερνοασφάλεια. Νομίζω ότι το, Συμβου... Κοινοβούλιο σε αυτές τις πολύ κουραστικές διαπραγματεύσεις έχει καταστήσει σαφές ότι εδώ δεν πρόκειται μόνο για αυτόν καθ' αυτόν τον οργανισμό αλλά γενικώ πώς μπορούμε να ε, εξασφαλίσουμε την κυβερνοασφάλεια στην κοινωνία μας. Δεν υπήρξε αντίθεση με την Κομισιόν και ε, ευχαριστώ την, ε, ε, την Επίτροπο που πραγματικά δεσμεύτηκε προσωπικά και θα ήθελα επίσης να ε, ευχαριστήσω και για την, τον κύριο Τσίζεστερ για την πολύ έξυπνη και με πολύ χιούμορ, με πολύ χιούμορ τρόπο που ε, χρησιμοποίησε για να ηγηθεί αυτή τη ε, όλη διαδικασία συζήτηση. Πραγματικά ο ΕΝΙΣ είναι ένα πολύ σημαντικό ε, οργανισμό έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει στον τομέα τη κυβερνοασφάλεια με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και γι' αυτό ευχαριστώ και του συναδέλφου που συμμετείχαν. Είναι πραγματικά ένα ακρογωνίο λίθο και νομίζω ότι με τούτο η συζήτηση αλλά και με την οδηγία για την για την κυβερνοασφάλεια. Έχουμε ένα πολύ καλό οπλοστάσιο και το χρειαζόμαστε έτσι ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Τικάω ένα λεπτό από τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε. Λαμβάνοντα υπόψη τη σημασία της ασφάλειας των δικτύων και των δεδομένων, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται έναν ισχυρό, σταθερό, μακροπρόθεσμα οργανισμό. Ως η εισηγητρία θεωρώ ότι σε ό,τι αφορά τον Ενίσα, τα πιο σημαντικά είναι τα άρθρα 2 και 3. Είναι τα άρθρα τα οποία θεσπίζουν ε, τους στόχους και την εντολή του οργανισμού. Διότι ο οργανισμός αυτός ε, έχει ευθύνη, θα έχει ευθύνη σε ό,τι αφορά την εφαρμογή όλων των νομικών διατάξεων που άπτονται της ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών. Θα πρέπει επίσης ο οργανισμός να συμβάλλει στην αύξηση των ε, δυνατοτήτων κρατών μελών να ανοιχνεύουν ενδεχόμενα προβλήματα ή κενά στα δίκτυα πληροφορικής. Επομένως, θα πρέπει ο οργανισμός να έχει έναν αυτόνομο επαρκή προπολογισμό και οι περισσότεροι υπάλληλοι θα πρέπει άμεσα να συμμετέχουν ε, στις εργασίες για την ε, υλοποίηση της αποστολής αυτού του οργανισμού. Δεν θα πρέπει να έχει μόνο 7 χρόνια ε, διάρκεια εντολή, πιστεύω. Θα πρέπει να έχει περισσότερα χρόνια. Ευχαριστώ. Εκ του Άλτε, τώρα, συνάδελφος Βαλεάν. Πρώτα απ' όλα θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή κύριο Τσίτσεστερ, γιατί πραγματικά ήταν ε, ε, πολύ αποφασισμένος ε, να υπάρξει συζήτηση για αυτή την έκθεση, έδειξε πείσμα, ισχυρογνωμοσύνη. Μετά από τρία χρόνια εντατικών διαπραγματεύσεων με Συμβούλιο και Επιτροπή πλέον θα ψηφίσουμε, πιστεύω, μια επιτυχημένη έκβαση. Δεν είναι συχνό το φαινόμενο, να αντιμετωπίζουμε τα πραγματικά ζητήματα, να αντιμετωπίζουμε τα πραγματικά πολιτικά ζητήματα πέρα από ταμπού, πέρα από συμφέροντα. Και ο κύριος Τσίτσεστερ κατάφερε μία έκθεση τετριμένη για απλά την παράταση της εντολής του ΕΝΙΖΑ ε, να μιλήσει για πραγματικά σημαντικά θέματα όπως είναι η διαφάνεια, η αποτελεσματική διαχείριση, η σχέση κόστος-οφέλους και είναι ορόσημο η έκθεση αυτή την καλωσορίζουμε, ιδίως ε, σε αυτούς τους καιρούς της κρίσης ε, που ε, έχουμε περιορισμό πόρων. Θα μας εμπνεύσει η εκθεσία του. Αυτό το νέο γραφείο συνδέσμου με βάση μέτρα την Αθήνα είναι ένα συμβιβασμό. Ελπίζουμε να προσελκύσει υψηλού επίπεδου ε, που θα να εργαστούν στον οργανισμό αυτό. Και με την ενισχυμένη του εντολή ο Νίσα μπορεί πλέον να τεδραματίσει το ρόλο του και να γίνει ένα σημαντικός εταίρος ε, στην προσπάθεια καταπολέμησης ε, του κοινωνικού και στην προσπάθεια να κατοχυρώσουμε την κυβερνοασφάλεια. Έχουμε κυβερνοαπειλές, ε, κυβερνοεπιθέσεις και στη ΣΥΠΑ βλέπουμε να αυξάνονται τα μέσα για την αντιμετώπιση τέτοιων απειλών. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι πραγματικά είναι υπαρκτός ο κίνδυνος και η απειλή αυτή. Ε, στον κυβερνοχώρο. Δεν θα πρέπει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αφήσει κατά μέρο αυτή την πρόκληση. Εμείς θέλουμε να έχουμε ένα οργανισμό, να έχουμε γενικά ευρωπαϊκούς οργανισμούς πιο ενισχυμένους και αποφασισμένους να δράσουν. Ευχαριστώ. Για τους πράσινους, η κυρία Άντας, τότε ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Τσίστερ, τον συγητή, και τους κύριους συγητές για τη βοήθεια που έκαναν και την κυρία Κρούς βέβαια για την δουλειά της στο ΕΝΙΣΑ. Πολλοί από, από μας μάθαμε πολλά πράγματα από τη δουλειά του ΕΝΙΣΑ που άλλωστε είναι εκεί για να συγκεντώνει πληροφορίες για τα δίκτυα και την ασφάλεια πληροφοριών. Τα μέτρα για το μέλλον θα πρέπει να είναι μέτρα που θα διευκολύνουν τη δουλειά του. Βεβαίω η ασφάλεια των δικτύων είναι πολιτικό τομέα και πρόσφατο πολιτικό τομέα. Ακόμα τώρα προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιο προστατεύεται και από ποιον. Προφανώ η Ενίζα έχει πολύ δραστηριότητα συλλογή πληροφοριών. Δεν ξέρω ωστόσο αν θα έπρεπε να αναθεωρήσουμε την κατάσταση. Τι ζητά το Κοινοβούλιο για την Ενίσα, τι θέλει να κάνει. Ευχαριστώ την Γκουε, ο Αγκουράκης. 1,5 λεπτό. Η αποπροσανατολιστική διαμάχη για το αν η έδρα του ΕΝΙΣΑ θα είναι στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην Αθήνα ή στη Χάγη επιχειρεί να συσκοτήσει ουσιαστικά ζητήματα. Η ουσία είναι η μετάλλαξη του οργανισμού και τα μεγάλα μονοπωλιακά συμφέροντα που συνδέονται με τον κυβερνοπόλεμο. Οι τροποποιήσει του κανονισμού που προτείνει η έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κινούνται σε ακόμα πιο αντιδραστική κατεύθυνση από την πρόταση τη Επιτροπή στην πραγματικότητα ο ενisa αντικαθίσταται από έναν άλλον οργανισμό στους σκοπούς του οποίου περιλαμβάνονται και αστυνομικά καθήκοντα όχι απλώς η ασφάλεια των δικτύων επικοινωνίας αλλά στην πραγματικότητα η αντιτρομοκρατική πολιτική της ευρωπαϊκής ένωσης και η καταπολέμηση τρομοκρατικών επιθέσεων στον κυβερνοχώρο η προστασία των υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας όπως λέγονται δημοσίων και ιδιωτικών έτσι ο οργανισμός αυτός προορίζεται να αποτελέσει την τεχνολογική υποδομή για τους κατασταλτικούς μηχανισμούς της ευρωπαϊκής ένωσης και των κρατών μελών ισοπεδώνοντας τα ανεπαρκή και ψευδεπίγραφα μέτρα δίθεν προστασίας προσωπικών δεδομένων στις εθνικές νομοθεσίες. θα συνδέεται άμεσα με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις κατασκευαστές εξοπλισμού δικτύων και αντίμετρων με τα ερευνητικά κέντρα και τα πανεπιστήμια. αποσκοπεί επίσης στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς και της ψηφιακής ατζέντα αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ. οι εξελίξεις με τον ενίσα είναι ακόμα μια απόδειξη για τον αντιλαϊκό χαρακτήρα της ευρωπαϊκής ένωσης που σαρώνει τα λαϊκά συμφέροντα τα δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες. γίνεται πιο επιτακτική ανάγκη της εργατικής λαϊκής πάλης για την ανατροπή της ευρωπαϊκής ένωσης για αποδέσμευση για κοινωνικοποιημένα μέσα παραγωγής. Ευχαριστώ οι υπόλοιποι Ο Τσουκαλάς, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Φοβούμαι ότι έχω διαφορετική γνώμη από τους συζητητές, μια που ούτε θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο ή η Επιτροπή στάθηκαν στο ύψος του στο θέμα του ΕΝΙΖΑ, ενός στρατηγικής σημασίας οργανισμού παρακολούθησα το θέμα του ενίζα πολύ στενά και ήταν φανερό ότι η πρώτη προτεραιότητα του εισηγητή κ. Τσίτσεστερ δεν ήταν η ισχυροποίηση του οργανισμού αλλά η μεταφορά της έδρας του από την κρήτη καταρχήν και από την ελλάδα κατά δεύτερον. επιστρατεύτηκαν κάθε είδους απίθανα επιχειρήματα ώστε να πιστούμε ότι η έδρα ενός τεχνολογικά προηγμένου οργανισμού που ασχολείται με την κυβερνοασφάλεια δεν μπορεί να βρίσκεται σε ένα ηλιόλουστο νησί του νότου προς αποκατάσταση τη τάξη θα ήθελα να πληροφορήσω του κύριου συναδέλφου ότι το νησί τη Κρήτη και το ηράκλειο αποτελούν σημείο επιστημονική και τεχνολογικής αριστεία πανευρωπαϊκής εμβέλεια. είναι προφανέ ότι η ενίζα θα έπρεπε να είναι ο οργανισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση που εξοχήν χρησιμοποιεί εργαλεία πληροφορική για να επιτελέσει το έργο του από οποιοδήποτε σημείο τη Ευρώπη. και δυστυχώς τα προηγούμενα χρόνια δόθηκε από την κυρία επίτροπο κάλυψη σε πρακτικέ διοίκηση και σε θλιβερά γεγονότα πίεση, ακόμη και απόλυση υπαλλήλων Καταδίκε από τον ευρωπαίο επόπτη Προστασία δεδομένων για παραβίες προσωπικών δεδομένων των υπαλλήλων του Ενίζα και καταδίκε του ευρωπαϊκού δικαστηρίου με ταυτόχρονη σπατάλη χρημάτων των ευρωπαίων πολιτών δεν πτώησαν την κυρία επίτροπο η οποία εξακολουθεί να στηρίζει τη διοίκηση κάτι που δεν θα γινόταν ανεκτό σε κανέναν άλλον οργανισμό. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, για τους παραπάνω λόγους προτίθεμαι να καταψηφίσω την πρόταση ανανέωσης της εντολής του οργανισμού. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βρούτσας. Ένα λεπτό. Δεν χρειάζεται να μιλήσω. Είναι προφανής ο σημαντικός ρόλος που θα παίξει και μελλοντικά δυστυχώ ο συμβιβασμό που δέχτηκε πρώτα απ' όλου η ελληνική κυβέρνηση μέσα σε περιβάλλον έντονων πιέσεων σχεδόν εκβιασμών θα έλεγα δύσκολα θα καταστήσει τον οργανισμό πιο αποτελεσματικό με παράλληλη λειτουργία σε δύο έδρε. είναι ένα συμβιβασμό που δεν αντανακλά τι θυσίε που έχει κάνει η ελλάδα μέσα σε συνθήκε πρωτοφανού οικονομική στενότητα που όλοι γνωρίζετε ώστε να κάνει το ηράκλειο έδρα κατάλληλη για τον ενίζα. για τον λόγο αυτό θέλω να καλέσω την επιτροπή να προβεί στα επόμενα χρόνια σε μια λεπτομερή αξιολόγηση της επιλογής της μεταφοράς της πλειοψηφίας του προσωπικού του οργανισμού στην αθήνα και σε μια ανάλυση του κόστους που θα προκύψει από αυτή τη μεταφορά καθώς και των προβλημάτων από την παράλληλη λειτουργία σε δύο έδρες. εδώ παλεύουμε να καταργήσουμε διπλές έδρες που έχουν αποδειχθεί κοστοβόρες και αναποτελεσματικές. αναρωτιέμαι λοιπόν ποιο μήνυμα στέλνουμε στους ευρωπαίους πολίτες σε περίοδο οικονομικής κρίσης. τέλος παρακαλώ την επιτροπή να έχει το θάρρος αν αντικειμενικά αποδειχθεί αυτή η κίνηση σπάταλη και υπονομευτική για τον οργανισμό να τη διορθώσει αμέσως. ευχαριστώ πολύ. Ο Κύριε ε. Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, τα δίκτυα και οι πληροφορίες και οι σχετικές υποδομές αλλά και η ασφάλειά τους σε όλο αυτό τον διαδικτυακό κόσμο που ζούμε είναι πραγματικά πολύ σημαντικά. Το κυβερνοέγκλημα είναι ένα πρόβλημα που αυξάνεται συνεχώς. Ε, το ε, ε, Ολλανδικό Ινστιτούτο έχει υπολογίσει ότι μόνο στη χώρα μου περίπου 10 δις ευρώ ετησίως καταβάλλονται για ζημίες. Και μάλιστα πρόσφατα είχαμε άλλο ένα πρόβλημα ε, από την τράπεζα ING. Ευτυχώς δεν υπήρξαν ε, απώλεια χρημάτων, αλλά πραγματικά αυτό κλονίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών σε αυτά τα συστήματα. Ο ΕΝΙΣ είναι ένα πολύ σημαντικό φορέα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δίκτυά μα πρέπει να είναι ισχυρά και ασφαλή. Μπορούμε να βελτιώσουμε τα πράγματα σε ό,τι αφορά την, ε, την εποπτεία από ευρωπαϊκή πλευρά. Βλέπουμε ότι υπάρχει αύξηση στο κυβερνό έγκλημα και όπω είπε και ο κύριο Έλερ, το κυβερνοέγκλημα και το σχετικό κέντρο για το κυβερνοέγκλημα μόλι άνοιξε στην ε, Europol, στη Χάγη. Δύο ερωτήματα λοιπόν. Ε, το επιπλέον κόστο ε, τη μεταγκατάσταση του ΕΝΗΣΑ είτε στην Αθήνα ποιο θα είναι, υπάρχουν χρήματα για να γίνει αυτό. Και επίση, για την αξιολόγηση στα πέντε χρόνια. Νομίζω ότι οι εξελίξει θα τρέξουν τόσο γρήγορα που σε τρία χρόνια θα πρέπει ήδη να δούμε τι γίνεται και ποια είναι η κατάσταση. Και ίσω να πρέπει το Κοινοβούλιο να το δει πολύ προσεκτικά αυτό. Νομίζω ότι το να, πάρουμε μόνο αυτό το, να κάνουμε μόνο αυτό το βήμα δεν αποτελεί εγγύηση. Ο κύριο Τσίτσεστερ βεβαίω προσπάθησε πάρα πολύ, έκανε πολύ καλή δουλειά και αυτό είναι καλό. Αλλά αναρωτιέμαι, έχουμε τα εργαλεία που χρειάζονται για, την, για τις νέες εξελίξεις που έρχονται. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κάλφιν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Καταρχάς, να εκφράσω την ικανοποίησή μου και τα συγχαρητήρια προς τον εισηγητή που κατάφερε και ολοκλήρωσε αυτό τον τρίλογο για τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Πιστεύω ότι είναι βέβαιο ότι η κυβερνοσφάλεια είναι θέμα του, του οποίου η σημασία αυξάνεται τελευταία χρόνια. Θα υπάρξει, δεν θα υπάρξει ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας αν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη και ανθεκτικότητα του συστήματος. Χρειαζόμαστε λοιπόν να δούμε το πλήρες ε, πλαίσιο και το, τη θεσμική δομή της ασφάλειας δικτύων στην Ευρώπη. Και χαίρο που υπάρχει πρόταση της Επιτροπής ήδη καθοδόν για τη στρατηγική κυβερνοασφάλισης και ε, ε, κυβερνοασφάλειας και μια σχετική οδηγία που θα εξετάσει το Κοινοβούλιο. Θα θέλω να δω μια πιο φιλόδοξη οδηγία για το ΕΝΙΣΑ. Να, μια οδηγία που θα επιτρέπει να έχει το ΕΝΙΖΑ μεγαλύτερη εντολή να δουλεύει περισσότερο από ότι στα θέματα εφαρμογής ε, θεμάτων κυβερνοασφάλειας. Αλλά και αυτό που έχουμε επιτάπητος είναι καλό αποτέλεσμα. Πρέπει να το ψηφίσουμε, να το υπερψηφίσουμε και να περιμένουμε τις εξέλιξεις. Ευχαριστώ. Η διαδικασία Catch the Eye. Ο κύριος Μικολάσικ, πρώτος ομιλητής. Πρόεδρε, το ίντερνετ το χρησιμοποιούν όλοι οι άνθρωποι όλων των, των ηλικιών και έχει προβλήματα ασφάλειας προφανώς. Υπάρχουν προγράμματα που μπορούν να περάσουν ως και συμπεριφέρονται ως η ανεπαρκής ε, προστασία επιτρέπει την διάδοση των ιών που επηρεάζει τη δουλειά των επιχειρήσεων και την ιδιωτική ζωή. Χρειάζεται λοιπόν να έχουμε ασφάλεια στο ίντερνετ και να μπορούν οι χρήστες να ξέρουν πώς θα, χρησιμοποιήσουν τα μέτρα αυτά. Πιστεύω ότι η ο οργανισμός είναι αναγκαίος, αλλά πρέπει να ξέρουμε τι εξουσίες θα έχει αυτός ο οργανισμός και τι θα κάνει τα αποτελέσματα. Με την οικονομική κρίση θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια και στο κόστος. Πιστεύω λοιπόν ότι το ενίσχυο θα πρέπει να έρθει στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Ευχαριστώ. Yeah. Ε, είναι, κεντρικό, είναι κεντρικό το θέμα για την ασφάλεια όλης της κοινωνίας μας. Στην τελευταία στρατηγική της ε, Επιτροπής για την Ασφάλεια ε, θα πρέπει κάθε κράτος να συμβάλλει στην ασφάλεια και την αποτροπή των ζημιών. Υπάρχει συντονισμό σε ευρωπαϊκό πλαίσιο για τον ΕΝΙΖΑ και μέσω της συνεργασίας αυτής θα φροντίσουμε ε, να καταπολεμήσουμε περισσότερο την, το κυβερνοέγκλημα ε, αναλαμβάνοντας δράση σε ενωσιακό επίπεδο και τώρα με τον κανονισμό γίνεται προσπάθεια να δημιουργηθεί οργανισμός που θα ανταποκρίνεται σε αυτές τις προκλήσεις. Δεν επιτρέπεται καθοριστικές υποδομές ε, να παραλύσουν που αφορούν πληρωμές κλπ. Σε αυτά τα πλαίσια χρειάζεται υψηλή ασφάλεια και για να εξυπηρετηθεί η οικονομία. Ο κ. Σέντσο, ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, να συγχαρώ καταρχήν τον κύριο Τσίτσεστερ και να χαιρετήσω τη συμφωνία που επετεύχθη για την παράταση της εντολής της, ε, του ΕΝΙΖΑ. Νομίζω ότι η ασφάλεια των δικτύων και των πληροφοριών πρέπει να είναι προτεραιότητα για όλη την Ένωση, δεδομένη της κοινωνικο οικονομική ζημιάς που απειλεί τα δίκτυα. Ο ΕΝΙΖΑ είναι ο μόνος οργανισμός που έχει την τεχνογνωσία για να εξασφαλίσει προστασία κατά των επιθέσεων και ο ρόλος και οι εξουσίες του πρέπει να αντικατοπτρίζουν αυτήν την πραγματικότητα. Είναι σημαντικό να μπορεί ο ΕΝΙΖΑ να στηρίζει τα, την ανάπτυξη των ε, δικτύων, των ΣΕΡΤ, που είναι αυτές οι ομάδες άμεση επέμβαση πληροφορικής που χρειάζονται σε επίπεδο ένωσης. Έχω πει πολύ συχνά ότι χρειάζεται σε ε, ευρωπαϊκό επίπεδο να έχουμε τα υψηλότερα πρότυπα ασφαλείας και ο ΕΝΙΖΑ μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο εδώ. Και ο κύριος ε, Πασκουά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Ο κανονισμός του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου ε, για τον ΕΝΙΖΑ δημιουργεί έναν οργανισμό ως προηγούμενο, ως διάδοχο του προηγούμενου στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο αυξανόμενο όγκο και η σημασία των ηλεκτρονικών επικοινωνιών αυξάνει την ανάγκη για ασφάλεια των πληροφοριών και των δικτύων και πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί ένα τέτοιο θεσμικό όργανο με μακρότερη εντολή από τα 5 με 7 χρόνια που προτείνονται. Ο, ε, συνεχείς ε, ε, αυτοσχεδιασμοί επηρέασαν αρνητικά την προηγούμενη περίοδο και τώρα θα γίνει μια αναθεώρηση των δραστηριοτήτων, έγινε μια αναθεώρηση των δραστηριοτήτων που τάσεται υπέρ σαφέστερων στόχων και πεδίου εφαρμογής του οργανισμού με αντίστοιχο προπολογισμό. Τα συστήματα συλλογής και ανάλυσης δεδομένων πρέπει να είναι στιβαρά για να μπορούν να αντιμετωπίζουν του συνεχώς ε, διαφοροποιούμενους ε, κινδύνους για την ασφάλεια. Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να προσεγγίσουμε το θέμα της μελλοντική εντολής του οργανισμού με τη μέγιστη δυνατή σοβαρότητα. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταία ομιλήτρια η κυρία Γκρέσλε. Κύριε Πρόεδρε, ως μέλος της ε, ε, διοργανικής ε, υπηρεσίας ε, χαιρετίζω αυτή την νομική βάση. Είναι ένα από τα πρώτα κείμενα τα οποία εκπονήθηκαν μετά από τη νέα συμφωνία που ήταν πολύ επώδυνη η δημιουργία της. Η υπηρεσία έχει μια έδρα στο Ηράκλειο και μια στην Αθήνα και θα ήθελα να συμβουλεύσω την Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να επιλέγονται οι ένδρες στο πλαίσιο του εφικτού και του λογικού ε, δεν είναι δυνατόν οι έδρε να αποτελέσουν, να ε, ε, δημιουργήσουν εμπόδια για την συντήρηση των υποδομών. Το να υπάρξει η έδρα τη υπηρεσία, το να δημιουργηθεί σε ένα νησί το οποίο είναι δυσπρόστο κατά τη διάρκεια του χειμώνα, ενώ υπάρχει μια άλλη έδρα στην Αθήνα, θεωρώ ότι δεν είναι λογικό και θα πρέπει να δημιουργηθούν οι προποθέσει ώστε η Επιτροπή να μπορεί να δουλεύει αξιόπιστα. Ευχαριστούμε πολύ κυρίες και κύριοι και τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στην Επίτροπο την κυρία Κρούς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Ε, Τέθηκαν κάποια ερωτηματικά εν σχέση με τις δύο έδρες της υπηρεσίας. Θα ήθελα να μιλήσω στα Ολλανδικά δεν θα πρέπει να υπάρχουν δύο οίκοι για... Ε, ε, ισχύει ότι υπάρχουν δύο σπίτια δημοκρατίας, ε, ένα στο Στρασβούργο και ένα στις Βρυξέλλες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μένα ούτως ή άλλως λειτουργεί σωστά το δίκτυο αυτό και όπως και το Κοινοβούλιο λειτουργεί σωστά παρόλο που υπάρχουν δύο έδρες. Τώρα, θα ήθελα να πω ότι ο κάθε μελητής σήμερα είπε ότι έχει συνείδηση της ε, σημασίας αυτής της υπηρεσίας και πολλοί βουλευτές ανέφεραν συγκεκριμένες ε, περιπτώσεις και πρόκειται για ένα ιδιαίτερο ευαίσθητο θέμα το οποίο θα πρέπει να προετοιμαστεί σωστά ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει εύρυθμα. Σήμερα είναι δυνατό να έχουμε ένα ασφαλές μέλλον για την ενίσα ούτε ώστε να μπορεί να πετύχει τους στόχους τους με τον πιο αποτελεσματικό δυνατό τρόπο. Και αυτό ήταν ε, το δικό σας ερώτημα που με απευθύνεται σε μια προηγούμενη συζήτηση. Πώς αποτελεσματικός μπορεί να είναι ο ΕΝΙΣΑ, ε, μιλώντας για την ίδια την οργάνωση, αλλά και τις σχέσεις κόστους ωφέλειας. Πώς ε, είναι δυνατόν να προσελκύσουμε τα πιο πρικισμένα άτομα του συνεργαστούν για, αυτή, για αυτόν τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό. Μία επικοδημητική συνεργασία μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Επιτροπής αυτή τη στιγμή γίνεται και ε, θεωρώ ότι είναι δυνατό και εύχομαι να υπάρξει ένα ευτυχές τέλος, μια ευτυχής έκβαση σε αυτή τη διαδικασία. Βεβαίω ορισμένοι έχουν κάποιους δισταγμούς και επιφυλάξεις γιατί υπάρχουν λίγα συγκεκριμένα δεδομένα και στοιχεία. Παρόλα αυτά, από την οικονομική άποψη, ε, αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει ένα επιχείρημα για να ταχθείτε κατά, γιατί μια έρευνα έχει αποδείξει ότι θα έχουμε ένα 50% ωφέλεια όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του ΕΝΙΖΑ και θα υπάρξουν οικονομίες 352.000 ευρώ ετησίως. Ε, και μιλάμε για 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό δεν σημαίνει μια κατάτμιση των πόρων γιατί αυτή τη στιγμή το μοντέλο βασίζεται σε μια ιδιαίτερως νοήμωνα προσέγγιση. Και δεν είναι η δική μου πρόταση. Πρόκειται για μια πρόταση ότι με την οργάνωση του ΟΝΙΖΑ έχει νόημα να διαμοιραστούν το λειτουργικό μέρος και το μέρος το οποίο σχετίζεται, συνδέεται με την έρευνα και την ε, λειτουργία της κεφαλής του ΕΝΙΖΑ. Ε, εν πάση περιπτώσει, ο ΕΝΙΖΑ πρόκειται να είναι ένας ε, είναι, ιδιαίτερος αποτελεσματικός οργανισμός. Είναι σημαντική η σύσταση αυτού του οργανισμού και είμαι ευγνώμων προς τον εισηγητή και τους ε, σκιώδεις. Ιδιαίτερα στον εισηγητή που ήταν παρόν εδώ, γιατί όλα αυτά δίνουν ε, τη δυνατότητα στον Ενίζα να λειτουργεί σωστά και στα χρονικά πλαίσια που έχουν προβλεφθεί. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Επίτροπη και τελειώνοντας θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Τσίτσεστερ. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τη συμβολή τους στη συζήτηση και ιδιαίτερως να ευχαριστήσω όσους ε, είπαν καλά λόγια και όσους ε, συμφώνησαν μαζί μου αλλά καταλαβαίνω και όσους ε, διαφωνούν. Θα ήθελα να τονίσω πως ε, η αναγνώριση του σοβαρότητας ε, του θέματος, ε, δηλαδή της ασφάλειας των δικτύων και των πληροφοριών, είναι και γι' αυτό και διοργανώθηκε αυτή η ακρόαση. Και κάναμε και μια νέα μελέτη, ο κύριος Πάσκο μίλησε για την μελέτη του 2004, κάναμε και μια νέα μελέτη που οδήγησε σε κάποια πορίσματα. Από την ακρόαση αυτό το οποίο εγώ αποκόμισα ήταν η σημασία της προσωπικής επαφής για τους κυβερνοεμπειρογνώμονες της, του οργανισμού. Οι βιντεοσυσκέψεις είναι πολύ ελκυστική ιδέα, αλλά ειλικρινά δεν υπάρχει αντικατάσταση, δεν υπάρχει υποκατάστατο για τη διαπροσωπική επαφή, ιδιαίτερα εκεί όπου πρέπει να διατηρηθεί η εμπιστοσύνη και η εμπιστευτικότητα στα θέματα ασφάλειας. Αυτό ήταν ένα πολύ σημαντικό μήνυμα που προέκυψε από την ακρόαση και από την μελέτη. Ε, θα πρέπει να σας πω ότι μας έδωσαν ε, έδωσε τροφή για σκέψη και δύο από αυτούς τις ε, τίτλους έλεγαν ότι η ευρωπαϊκή, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα κινδυνεύουν. Δύο διαφορετικά παραδείγματα μας ε, αναφέρθηκαν, ότι δηλαδή δεν είναι άτρωτα τα θεσμικά όργανα. δόθηκαν 12 συστάσεις, από τις οποίες 8 έγιναν δεκτές και ενσωματώθηκαν στο κείμενο. Και εκεί συμπεριλαμβανόταν η εγκατάσταση του υπηρεσία αυτή στην Αθήνα και μία-δυο έμειναν εκτός και κάποιες σε, σε κρεμότητα. Το θέμα ήταν ότι διαρκώ δική μα μέρημνα ήταν αυτή η υπηρεσία, αυτό ο οργανισμό να είναι πιο αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που υπάρχουν και αυτών που δεν γνωρίζουμε ακόμα για το μέλλον. Και ελπίζω ότι δώσαμε το νομοθετικό πλαίσιο στο οργανισμό αυτό να προχωρήσει ε, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώνεται η συζήτηση και η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 12. Let's continue with point of our... Συνεχίζουμε με το επόμενο σημείο της ημερής.